Jeg Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα στα δανέζικα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Σας ενθαρρύνω να το πράξετε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών και βλέπω ότι από τα 24 μέλη μόνο 6 είναι από πριν, από το προηγούμενο κοινοβούλιο. Άρα θα χρειαστεί πολύ σύντομα να μάθετε πολλά πράγματα. Για την Επιτροπή Αναφορών θα πω ότι πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή επιτροπή, συναρπαστική, εφόσον έρεται στο ύψος των προσδοκιών των πολιτών μας. Είμαστε μια επιτροπή η οποία δεν εξετάζει τα κομματικά ή εθνικά συμφέροντα. Η Επιτροπή μας οφείλει να είναι αξιόπιστη διότι είναι Επιτροπή Αναφορών των Πολιτών. Επιθυμώ να σας ενθαρρύνω όλες και όλους στη δουλειά μας και σήμερα και στα χρόνια που έρχονται, γιατί η Επιτροπή Αναφορών είναι το πρόσωπο του Κοινοβουλίου απέναντι στους πολίτες. Πολύ σημαντική λοιπόν για τη στήριξη της νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου. Τώρα, έχουν καταχωριστεί όλες και όλοι οι παρόντες και γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν βάλει τις κάρτες τους, ό,τι θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε, αρκεί να ψηφίσετε. Λοιπόν, βάλτε τις κάρτες σας στην ε, σχισμή να δούμε ότι όντως όλες οι πολιτικές ομάδες, ψηφίστε οτιδήποτε θέλετε, πατήστε κάποιο κουμπί, όποιο κουμπί θέλετε, μπροστά σας είναι τα ισχυσμοί με τα κουμπιά, ό,τι θέλετε. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πατήστε λοιπόν κάποιο κουμπί για να δούμε ότι καταχωρείται η παρουσία σας. Χρειαζόμαστε λοιπόν 10 μέλη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουμε 10 μέλη του Λαϊκού Κόμματος, 9 από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, 3 μέλη από την ε, πολιτική ομάδα ECR, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, 3 από τους Ελευθέρους, ALDE, 3 από την Ενωτική Αριστερά, 3 από τους Πράσινους, δύο από την ομάδα EFDD και έναν μη εγγεγραμμένο. Είναι σωστό, βγαίνει το άθροισμα. Κάποιος ή κάποια δεν έχει την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας. Έχει καλώς. Πρώτα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκλογή Προέδρου. Θα ήθελα να ακούσω ποιος είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Επιτροπής Αναφορών. Όνομά σας. Προτείνω την Eleanor Ήβη. Άλλες ε, προτάσεις. Εσείς. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία Σεσίλια Βίκστρομ. Ε, Η προεδρεύουσα κυρία Άουκεν. Δέχονται και οι δύο υποψήφιες. Έχει καλώς, ευχαριστώ. Άρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, κάποιος διακόπτει. Δεν διεξάγεται συζήτηση, δεν προβλέπεται να διεξαχθεί συζήτηση. Αλλά σας παρακαλώ να δεχτείτε, παρακαλώ την Επιτροπή να δεχθεί μια τοποθέτηση δύο λεπτών από κάθε υποψήφια. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Ε, είμαι υποψήφια για αυτή την επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω από εσά συναδέλφου ε, αν θεωρείτε ότι ο ρόλο μα ω Ευρωβουλευτών είναι ένα επάγγελμα ή αν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε στου πολίτε. Εγώ εκλέγομαι από το δίκτυο με μια νέα και δημοκρατική μέθοδο μέσω online εκλογών ή το αποτέλεσμα μια, ενός πολιτικού πειράματος διεθνούς ελληνικούς και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Είμαι λοιπόν μια πολίτης στην υπηρεσία των πολιτών και για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα αλλά αποστολή. Μετά από τις σημερινές ψηφοφορίες που έγιναν ε, ε, όλη την ημέρα, θα ήθελα να καταγγείλω ενώπιον όλων σας πως σήμερα παραβιάστηκε η μέθοδος ε, DONT που εγγυάται την κατάλληλη αντιπροσωπευτικότητα σε θεσμικό επίπεδο εκείνων των μειονοτικών ομάδων που έχουν όμως νόμιμα εκλεγεί από εκατομμύρια πολίτες, όπως το κίνημα των πέντε αστέρων στην Ιταλία εναλλακτικά ανταγωνιστικές ομάδες έχουν, έχουν ενωθεί για να εμποδίσουν τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου DONT, για να εμποδίσουν ε, τις, ε, για να, αναλάβουν μάλλον τι προεδρίες και τι αντιπροεδρίες σε όλες τις επιτροπές. Εγώ μιλώ εξ ονόματό μου και εξ ονόματο τη ομάδα μου και του κινήματος των πέντε αστέρων. Είμαι πραγματικά εξοργισμένη απέναντι σε αυτή τη δράση που θεωρώ αντιδημοκρατική και ανήθικη και που στηρίζει ένα ολιγαρχικό σύστημα αυτοπροστασία και αυτοσυνέχισης, αυτοδιατήρησης γιατί τιμωρηθήκαμε, για ποιους λόγους, θα ήθελα να έχω μια απάντηση από εσά. Η σημερινή ψηφοφορία από ένα βήμα πίσω για τη δημοκρατία. Με την ελπίδα πως αυτό δεν θα γίνει στο μέλλον, η ομάδα EFD και το κίνημα 5 αστέρων θα είμαστε εδώ και θα επαγρυπνούμε ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. η Πρόεδρος. Σισίλια Βέξτρομ, θέλετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι υπερήφανη και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι υποψηφία για την ανάληψη του αξιώματος της Προέδρου αυτή της τόσο σημαντικής για τους Ευρωπαίους πολίτες Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν θέλω να προβώ σε δήλωση υποσχέσεων. Ένα μόνο πράγμα θα πω, ότι θα είμαι ειλικρινής και τίμια πρόεδρος, διαμεσολαβήτρια για όλους και όλες τους βουλευτές. Σκοπός μου είναι να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα όπου όλοι θα έχουν την διάθεση να τοποθετούνται ελεύθερα και να αναπτύσσεται μια συζήτηση μεταξύ μας ως πολιτικών, ανδρών και γυναικών, εκλεγμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πράξω λοιπόν κάθε τι που είναι στις δυνάμεις μου, θα ακούω και θα μιλώ με όλους και όλες τις συναδέλφους μου από όλα τα κόμματα. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Βέγκστρομ. Πριν προχωρήσουμε στην διεξαγωγή της ψηφοφορίας, έχουμε αναπληρωματικό μέλος από την Ενωτική Αριστερά. Τώρα θα προσπαθήσω να προφέρω τα ονόματα. Μέρι Νελπιόνε από την Γκουε, η οποία αντικαθίσταται από την κυρία Αντζέλικα Μπεντίνα. Η κυρία Σοφία Σακοράφα εκπροσωπείται από την Άνια Χάσελκαμπ. Και ο Τάκης Χατζηγεωργίου εκπροσωπείται από την κυρία Λόπες. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Μαλένη Μίτση εκπροσωπείται από την κυρία Ντάλη και από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κ. Βοητσεχόφσκι αντικαθιστά τον κύριο Χάνεν. Καλά λοιπόν, αφού πέρασα και αυτό και αυτή τη δοκιμασία, ας αρχίσω με τα αγγλικά τώρα όσοι ψηφίζουν, όσε και όσοι ψηφίζουν υπέρ τη κυρία Εύη θα ψηφίσουν πράσινο, θα πατήσουν πράσινο. Υπέρ τη κυρία Βέγστρομ κόκκινο κουμπί. Και αρχίζει η ψηφοφορία ευθύ αμέσω. Θα επαναλάβω, θα επαναλάβω καλύτερα. Όπως ε, προβλέπει και η συμφωνία που έγινε νομίζω στην διάσκεψη πρώην πολιτικών ομάδων, η ψηφοφορία θα γίνει ω εξή όσες και όσοι ψηφίζουν την κυρία Εύη πατούν το πράσινο κουμπί. Όσες και όσοι ψηφίζουν την κυρία Βέξτρομ πατούν το κόκκινο κουμπί. Τώρα είναι κατανοητό αυτό που είπα. Καταλάβατε όλοι. Με συγχωρείτε. Στη μετάφραση κάπως ε, μου τα μπερδέψανε, λέει μια βουλευτής. Να το πω τι στα γερμανικά, λέει και Τώρα είναι κατανοητά τα όσα είπα. Είναι σαφή. Καλά λοιπόν. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Μένουν ακόμα πέντε να ψηφίσουν. Has everybody voted now? Ψηφίσατε όλες και όλοι. Υπάρχει Κάποιος που δεν ψήφισε. Ωραία, τότε κλείνει η ψηφοφορία, λίγη. Βλέπετε λοιπόν τα νούμερα, το αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι η κυρία Βίξτρομ εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής Αναφόρων. Μπορείτε να έρθετε εδώ παρακαλώ. Yeah, Thank you very much. Thank... Η κυρία Βίξτρομ, νέα πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Προς την κυρία Εύη απευθύνω. Είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε μαζί να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα καλή συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμού. Αυτό είναι ο στόχο μου στην ανάληψη των καθηκόντων μου, να συνεργαστώ στενά με όλε και όλου σα, ανεξαρτήτω προορισμού σα, ε, συγγνώμη, ανεξαρτήτω προελεύσεώ σα και ανεξαρτήτως συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε πολιτική ομάδα. Όπως είπα θέλω να είμαι πρόεδρος που θα σέβεται όλες και όλους και στην παρούσα επιτροπή που είναι ιδιαίτερη όπως είπε και η κυρία Άουκεν προηγουμένως μπορούμε όντως να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με στόχο να φτιάξουμε γέφυρες προς τους πολίτες και των 28 χωρών μελών μας, γιατί χρειάζονται αυτές οι γέφυρες. Να συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε υπέρ των αγαθών στόχων που ε, για αυτούς έχει φτιαχτεί η Επιτροπή Αναφόρων. Είμαι συγκινημένη όπως αντιλαμβάνεστε και είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς την ε, κατεύθυνση της επίτευξης καλών αποτελεσμάτων. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη δουλειά μας. Μια φορά όσοι δεν έχουμε μητρική γλώσσα τα αγγλικά, είναι χρήσιμο να τα μιλούμε ωστόσο, έστω και αν δεν μπορούμε τόσο καλά, γιατί τότε δεν θα χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή τη μετάφραση. Τώρα η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την έννοια ότι θα προχωρήσουμε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων και παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις υποψηφιότητες. Είμαι ο κ. Άκερ. Προτείνω την Ελεονόρα Εύη. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Πρώτον, σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Θα είναι θαυμάσια συνεργασία μαζί σας, είμαι βέβαιος. Για πρώτη αντιπροεδρία, το Λαϊκό Κόμμα προτείνει την κυρία Φέραγκουτ. Εστέρας Φαραγκούτ. Φέραγκούτ μάλλον πιο σωστό. Άλλες προτάσεις, άλλες υποψηφιότητες. So it's green for this Άρα λοιπόν, πράσινο για την κυρία Εύη, κόκκινο κουμπί για την κυρία Εστάρα Σφεραγκούτ. Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. τώρα να κλείσουμε λοιπόν. Μάλιστα, τα αποτελέσματα. Δέκα ψήφι υπέρ, λέει η πρόεδρος, υπέρ της κυρίας εννοεί, και 20 υπέρ της κυρίας Εστάλας Φεραγκούτ. Έτσι λοιπόν, συγχαρητήρια και ελάτε παρακαλώ να καθίσετε δίπλα μου. now we need to... Τώρα να ψηφίσουμε την δεύτερη αντιπροεδρία. Εσείς κύριε Γιάρ. Εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος προτείνω την υποψηφιότητα την κυρία Ρομπέρτα Μιτζούλα. Mr. Eka. Uh, I propose Προτείνω την Eleanor Evie. Ωραία λοιπόν. Πράσινο για την κυρία Μετζόλα και κόκκινο για την κυρία Εύη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Έδειξε η ψηφοφορία. 20 λοιπόν ψήφι υπέρ της κυρίας Μεζόλα και 11 για την ε, υπέρ της κυρίας Εύη. Η κυρία Μετσόλα λοιπόν είναι παρούσα, δεν είναι παρούσα. Να προχωρήσουμε τότε στην ε, τρίτη υποψηφιότητα. υποψηφιότητες εσείς. Μαρλέν Μισή εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Άλλες υποψηφιότητες. Ο κύριος Άκερ επιμένει στην κυρία Ελεονόρα Εύη. Τι έκπληξη. Πράσινο η κυρία Μίτση και κόκκινο η κυρία Εύη. Αρχίζει η φοφορία. έληξε η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως και για την προηγούμενη. Θα προχωρήσουμε τότε... Α, πρώτα υποψηφιότητες. Κύριε Άκερ. Ναι, ναι, εντάξει, κυρία Εύη, ναι, ναι. Και, κύριε Γιάρ. Η κυρία Άουκεν ε, αστείευεται χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Γιάρ, εσείς. το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν φταίει στο κάτω της γραφής που μας προτίμησαν οι υποψηφοφόροι. Προτείνουμε στην τέταρτη διπροεδρία τον κύριο Παουλτσάκη. Ευχαριστώ κύριε Γιά. Είναι και άλλες υποψηφιότητες. σχόλιο κυρία Για πρώτη φορά βλέπω να μην ακολουθούμε τα ιωθώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να είμαστε αντίθετοι με κάποια υποψήφια, αλλά να βρισκόμαστε αντιμέτωποι, να στεκόμαστε απέναντι σε μια πολιτική ομάδα, έστω και αν ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις, βλέπω τι γίνεται Λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εμεί είμαστε οι περισσότεροι, έχουμε την πλειοψηφία. Θα κάνετε ό,τι λέμε. Ελπίζω ότι είναι η τελευταία φορά που ακούω σε αυτήν εδώ την Επιτροπή αυτό το επιχείρημα. Ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχει και άλλος κανείς ε, την επιθυμία να ομιλήσει. Έχετε το λόγο. Θέλω εκ μέρους του ECR να επισημάνω ότι και σε άλλες δύο επιτροπές είδαμε προηγουμένως υποψήφιος και υποψήφια από το κίνημα των πέντε αστέρων να αποκλείονται παρά την μέθοδο DONT η οποία έχει αποφαστεί ότι ισχύει. Και ξαφνικά βλέπουμε εδώ να επιμένουν οι συνάδελφοι στην απόρριψη της υποψηφιότητας της κυρίας Ήβη και τώρα άκουσα τον συνάδελφο από το Λαϊκό Κόμμα να λέει και να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μέθοδος don't. Λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς είμαστε αντίθετοι στον οποιοδήποτε αποκλεισμό πολιτικής ομάδας, διαφωνούμε μαζί τους, αλλά είμαστε αντίθετοι στις διαδικασίες που γίνονται και αποκλείονται ειδικότερα οι υποψήφοι του κινήματος των πέντε αστέρων. Και αυτό θέλουμε να το επισημάνουμε. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you. Σας ευχαριστώ για την δήλωσή σας. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο υποψηφιότητες, Πολ Ζάκη, πράσινο κουμπί και πάλι κόκκινο για την κυρία Ήβη. Αρχίζει η ψηφοφορία.